So, meine Damen und Herren, liebe... Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε την συνεδρίαση με τις ψηφοφορίες. Πριν όμως προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες, έχω μία ανακοίνωση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μου ανακοίνωσαν ότι διορίζεται στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ο κ. Γκονζάλες Πόνς αντι, αντικαθιστώντας τον κύριο Ιτουργκάης. Υπάρχουν ενστάσεις. Όχι. Άρα ο διορισμός ε, του προαναφερθέντος συναδέλφου ισχύει. Προχωρώ στην ψηφοφορία για το πρόγραμμα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016. Κοινό ψήφισμα